έχουν ήδη πετύχει αρκετά πράγματα και ο διάλογος έχει καρποφορήσει για τον περιορισμό της τρομοκρατίας στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μονίθ και έτσι εδώ ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις ενός λεπτού. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση τη κυρία Ντεκάισερ για συστήματα υγειονομική περίθλιψης στην υποσοχάρη Αφρική και παγκόσμια υγεία. Παρακαλώ. Για τέσσερα λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε ακόμα μεταξύ μας. Η έκθεση αυτή απαντά ε, κατά κάποιο τρόπο σε μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, υγεία σε ολοκληρωμένο επίπεδο, αλλά θέλει να δει τα πράγματα από μια ιδιαίτερη οπτική ε, γωνία ε, και να ασχοληθεί περισσότερο με τα προγράμματα αλληλασφάλισης υγείας που ανθούν αυτή τη στιγμή στην Αφρική η κατάσταση της υγείας στην ε, ε, Αφρική αυτή τη στιγμή είναι δραματική παρά τη βοήθεια διεθνών ε, οργανισμών και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους. Κλιματική αλλαγή, χρηματοπιστωτική κρίση, πόλεμοι, κακή διακυβέρνηση σε πολλές χώρες ευθόνος ε, λόγω των ε, ε, εξωτερικών παραγόντων, λόγω της, του πλούτου που βρίσκουμε στην Αφρική και επομένως ασθένειες όπως η ελονοσία, εφηματίωση και άλλες έχουν αρχίσει να ανθίζουν εκ νέου. Θα ήθελα εδώ να χαιρετήσω την εργασία και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και κάποιων εκκλησιών που κάνουν πραγματικά αξιοθαύμαστη και αξιοπρόσεκτη εργασία σε απομακρυσμένες περιοχές, σε εμπόλεμες ζώνες κλπ. Ε, υπάρχουν τα λεγόμενα κάθετα ταμεία ε, τα οποία θέλουν να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα υγείας όπως ελονοσία, AIDS κλπ. Ε, τα ταμεία αυτά απορροφούν πάρα πολλά χρήματα, είναι ελκυστικά για τους δωρητές αλλά στην ουσία αυτά τα ταμεία τα οποία επιτυγχάνουν το στόχο τους τελικά καλύπτουν μονάχα ένα τμήμα του προβλήματος γιατί ε, πεθαίνουν ε, αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερα παιδιά λόγω έλλειψης ε, πόσιμου νερού παρά από το AIDS ή από την ειρηνοσία. Επομένως, επομένως από την αρχή της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν κάποιες πρωτοβουλίες για προγράμματα ασφάλισης, κυρίως δε αλληλασφάλισης υγείας, Mutuel Αυτά τα συστήματα λοιπόν ε, της αλληλασφάλισης υγείας θέλουν ε, να ε, να δημιουργήσουν ένα γενικότερο πλαίσιο για την κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης σε πρόσβαση σε φάρμακα σε συνδυασμό με διάφορα ταμεία έτσι ώστε να υπάρξει διασφαλισμένη κάλυψη περίθελψης υγείας και πρόσβασης σε φάρμακα ε, και βεβαίως ε, συνδυασμένη με μια νέα κοινωνική ε, δυναμική. Ε, υπάρχουν λοιπόν διάφορες MTL, διάφορα προγράμματα αλληλασφάλισης, αλληλασφάλισης ε, μικρών ταμείων, γυναικών κτλ. Ε, και βεβαίως το σημαντικό είναι αυτό το σύστημα των δομών αλληλασφάλισης να είναι καλά συντονισμένα μεταξύ τους. Εάν μπορούν να δημιουργηθούν και να υπάρξουν αυτές οι δομές αλληλασφάλισης μπορούν να υπάρξουν μονάχα μέσα από οριζόντια συστήματα. Δηλαδή γιατί κανείς να πάει να ε, πληρώσει ας πούμε για να ασφαλιστεί ε, ε, απέναντι για, ενδεχόμενο ας πούμε εγχείρηση εάν δεν υπάρχει δυνατότητα εγχείρηση γιατί κοντά στο μέρος που ζει κανείς δεν υπάρχει καθόλου νοσοκομείο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να βρεθούν νέα συστήματα τα οποία θα ε, προωθήσουν τα οριζόντια ε, συστήματα έστω και αν πρέπει να ζητήσουμε από τα κάθετα συστήματα υγείας να βοηθήσουν αυτά τα οριζόντια συστήματα. Αυτή είναι η έννοια της έκθεσής μου. Βλέπω ότι δεν έχω χρόνο αλλά ενδεχομένως ε, εάν κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να ρωτήσουν κάτι συγκεκριμένα για την αναπαραγωγική υγεία που αναφέρεται στο, στην έκθεσή μου βεβαίως έχω κάθε διάθεση να απαντήσω. Για το Catch the Eye, ένας έχει ζητήσει μόνο το λόγο. Α, τρεις, διορθώνει ο πρόεδρος. Ο κύριος Ρινάλντι πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Ντικεζέρ τα είπε σχεδόν όλα. Ε, εγώ θα ήθελα το λεπτό μου να, στο λεπτό μου να αναφερθώ σε ένα παιδί που γνώρισα στη Λουάντα, στην ε, Αγγόλα, όταν είμαστε εκεί για τις εργασίες ε, ε, της Ισομερούς Συνελεύσεως το τέλη του 2009 είναι ήταν ένα παιδί το οποίο πέθαινε λόγω ασιτίας και πέθανε ακριβώς δίπλα ε, στο μέρος που εμείς συναντιόμαστε και δίπλα στο μεγάλο ε, γήπεδο στο οποίο θα πεζόντουσαν μετά αγώνες του παγκόσμιου ε, κυπέλου. Είδα λοιπόν αυτό αλλά και άλλα παιδιά να πεθαίνουν, να υποφέρουν στην αγκαλιά των μανάδων τους <coughs> λόγω ασυτείας. Πιστεύουμε ότι είναι αμαρτία ένα τέτοιο θέαμα ε, είναι αμαρτία και καταδεικνύει σαφώς την αποτυχία των συστημάτων μας. και νομίζουμε ότι και στην Αγγόλα ε, ε, καταδεικνύει σαφώς και την, τον κακό καταμερισμό του πλούτου. Ευχαριστούμε πολύ για την μαρτυρία αυτή. Η κυρία Μπόσκα έχει τώρα το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Παρά κάποιες, τις κάποιες επιφυλάξεις που έχω εναντί αυτής της έκθεσης, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ντεκάιζερ. Έχει δείξει, όπως και πολλές φορές στο παρελθόν, πως γνωρίζει τις ε, πολιτικές ε, τις αναπτυξιακές και δεν είναι αδιάφορες στις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων. Στην υποσαχάρια Αφρική το επίπεδο ιατρικής περίθλιψης είναι πραγματικά πολύ κακό. Λυπούμε για το ότι κάποιες τροπολογίες δεν έγιναν δεκτέν, δεκτές. Κάποιες τροπολογίες που κατέθεσα συχνά μιλάμε για έγγραφα των διασκέψεων του Καΐρου και του Πεκίνου και δεν γίνονται δεκτές οι παραπομπές μου γιατί κάποιοι συνάδελφοι θεωρούν πως κάποιες παράγραφοι δεν αφορούν ε, το θέμα της αναπαραγωγικής υγείας στην Ευρώπη. Δεν θέμε να σεβαστούμε τις ε, τοπικές ε, ιδιαιτερότητες των κρατών στην υποσαχάρια Αφρική και έτσι μόνο θα χειροτερεύσει η υγεία των ανθρώπων. Ευχαριστώ, κ. Νικολάζικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνωρίζει την υγεία βεβαίως ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Εγώ προσωπικά θεωρώ πως το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα με το δικαίωμα στην ζωή. Έχουν συγκεκριμένο νόημα αυτά τα δικαιώματα στην υποσαχάρια Αφρική. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα την υπεύθυνη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην υγεία στην υποσαχάρια Αφρική. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθεί την έκτρωση ως ε, δικαίωμα γιατί το λεγόμενο αυτό δικαίωμα δεν αναφέρεται πουθενά σε διεθνείς συνθήκες. Αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί την ζωή μητέρων με τα παιδιά τους, να διευκολύνει τη ζωή τους και να βρει τρόπους να προστατεύσει τη ζωή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της δεν έχουν ρήτρε στις ε, Εμπορικέ συνθήκες που θα επιτρέψουν σε ανθρώπους να λάβουν βασικά φάρμακα. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη θνησιμότητα σε αυτές τις χώρες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Φιλίπκας δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να σας υποβάλω κάποια σχόλια και σκέψεις. Για να σας πω μάλιστα την αλήθεια, Πάντα η Επιτροπή βέβαια είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου και εγώ πολύ χαίρομαι που άκουσα και την κυρία Ντεκάιζερ και τους άλλους για ένα θέμα το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει πολύ. Η κυρία, Ντεκάιζερ ως ε, επίτροπος και πέρα από τις δραστηριότητε μου στον οικονομικό τομέα μετά από τις επισκέψεις που έκανα στις διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ξέρετε ότι τα θέματα που συζητάμε στο νομικό τομέα είναι διατλαντικά, πήγα και στην Αντίση Σαβέβα, τέλη Ιουλίου, για να συναντηθώ με ηγέτες της Αφρικανικής Ένωσης, γιατί εδώ και χρόνια ζητάω μια νέα ε, πολιτική εταιρική σχέση με την Αφρικανική Ήπειρο. Σίγουρα υπάρχουν θέματα που συνδέονται με την κρίση και που αντικατοπτρίζονται στη δικιά σας παρέμβαση, η κατάσταση στις αγορές, η καταπολέμηση ε, του, της νομιμοποίησης του παράνομου χρήματος, η οικονομική διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της κερδοσκοπίας ε, για τις πρώτες ύλες, από τις οποίες εξαρτάται η Αφρική τρόφιμα. Αποφάσισα λοιπόν, μετά από τη συνάντηση αυτή, αποφάσισα με τους συναδέλφους να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Σας συγχαρώ και εκ μέρους του κύριου Πίλκας και εκ μέρους μου για την τόσο καλή εκθεσή σας. Εσείς αναφέρεστε στην κατάσταση της υγείας στις υπονάπτυξη χώρες και δεν μιλάμε μόνο για την Αφρική. ήμουν στην Αιτή πριν από μερικές εβδομάδες. Μετά από την κυρία Άστον και την κυρία Τζόρτζεβα που πήγαν εκεί τον κύριο Πίβαλς, πήγα και εγώ. Και βλέπουμε ότι και σε τέτοιες χώρες υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την υγεία. Όπως λέει και ο κύριος Ρινάλντι, το γεγονός ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι πρόωρα χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις υποανάπτυξη χώρες για λόγους που έχουν γιατριά και θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί με τα χρήματα που ξοδεύουμε στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα κατοικίδια μας ζώα. 2% των στρατιωτικών δαπανών παγκοσμίω επίσης θα φτάνανε. Λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση είναι απαράδεκτη. Οι κοινωνικές πολιτικές, βιώσιμες κοινωνικές πολιτικές και υπέρ της υγείας θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα των χωρών για να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η υγεία είναι δικαίωμα για όλους. Επιπλέον αποτελεί και μέρος της οικονομικής ανάπτυξης. Θέλουμε συστήματα υγείας που να ε, βασίζονται σε λιγότερο από 30 ευρώ κατά το χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε διαθεσιμότητα φαρμάκων έτσι όπως χρειάζονται και ιατρικό προσωπικό έτσι όπως χρειαζόμαστε. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω εκ μέρους του κύριου Πίλουκας είναι ότι θα επιμείνουμε ώστε να τιμήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθήσει την ανάπτυξη των τρίτων χωρών εκείνων που τη χρειάζονται περισσότερο. Το θέμα της υγείας είναι προτεραιότητα για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Θέλουμε λοιπόν πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες για να βελτιωθεί η υγεία την κυρία Ζαρμπόφσκα τώρα, θέλω να πω ότι τρίτες χώρες που όμως δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια κατάσταση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από χώρα σε χώρα. μεταξύ των υπονάπτυξη των λιγότερων αναπτυγμένων της Αφρικής. Θέλουμε πάντως η Επιτροπή να συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές προσπάθειες που γίνονται για να καταπολεμηθούν διάφορες ασθένειες όπως είναι η φυματίωση, το AIDS κλπ. Ελονοσία, πολυμελίτητα κλπ. Βοηθούν οι μη κυβερνικέ οργανώσει. Στην ΑΕΤ πριν από λίγε μέρε ήμουν και είδα πόσο αποφασιστικό ρόλο έχουν για να βοηθήσουν και για να βοηθήσουν να δαπανηθούν καλά τα χρήματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων δωρητών. Χρειάζονται λοιπόν συγκεκριμένα αποτελέσματα και στην Ευρώπη και στις υποανάπτυξη λοιπόν, χώρες. Τώρα να μιλάμε απλώς για το επίπεδο των πόρων, αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχει κάποια συνοχή στις πολιτικές μας για την μετανάστευση, για τους επαγγελματίες υγείας ή για το εμπόριο φαρμάκων. Χρειάζεται λοιπόν μια σφαιρική συμφωνία η οποία να βοηθάει και αν μη τι άλλο να μην βλάπτει αυτού που περισσότερο έχουν ανάγκη από τέτοιε πολιτικές στον κόσμο. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες, δύο πράγματα θέλω να σας πω κύριε Δικάιζερ που σας ενδιαφέρουν πιστεύω. Το ένα έχει κάνει για το Single Market Act. Εγώ σκοπεύω να ευνοήσω και να ενθαρρύνω του τομεί εκείνους που μπορούν να βοηθήσουν. Τις δομέ εκείνες, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και να διευκολύνω τη δουλειά τους προ όφελο των πιο φτωχών χωρών. Υπάρχει και ένα δεύτερο πράγμα το οποίο με απασχολεί πολύ που είναι το θέμα της παραποίησης προϊόντων, των πλαστών προϊόντων. Στο σχέδιο που θα σας παρουσιάσω τον επόμενο φθινόπορο για την καταπολέμηση της πειρατείας και των πλαστών προϊόντων έχω ένα κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της τεχνολογίας που εντοπίζει τέτοια προϊόντα, που ανοιχνεύει τέτοια προϊόντα, όπως επίσης και για την κατάρτιση των ειδικών στα τελωνία και αλλού για να εντοπίζουν τέτοια προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν και ένα κεφάλαιο για συνεργασία με τις χώρες από τις οποίες μας έρχονται τα πλαστά προϊόντα, αλλά και για τις χώρες όπου προκαλείται μεγαλύτερη ζημιά εξαιτίας αυτών των ε, πλαστών προϊόντων. Βάσει της ανάλυσης λοιπόν που σας και γράφησα, η Ένωση έχει καταλήξει σε μέτρα για την υγεία και όπως είπα, οι πόροι για την ε, ανάπτυξη δεν αρκούν. Βάσει της ανάλυσής σας, της έκθεσής σας, πολύ σωστά φαίνεται αυτό. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να ενισχύσουμε τα συστήματα χρηματοδότησης. Δεν είναι τέλεια και δεν υπάρχει και καμία τέλεια λύση για όλους. Χρειάζεται ένα σύστημα ασφάλισης που να βασίζεται σε ιδιωτικά συστήματα, αλλά και αυτό δεν φτάνει για να υπάρξει δίκαια και συνολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για χρηματοδότηση συστημάτων υγείας και να διέπονται από ισότητα. Συστήματα στα οποία να μπορούν όλοι να συμμετέχουν. Ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεισφορά του, για την ε, αλληλεγγύη προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις.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 Καλό βράδυ σε όλους. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να πω, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχει μερική διάταξη και είναι στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.